Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι, οπότε η προτινόμενη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι ακριβώς ε, η δήλωση της ΕΕ εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Στην συζήτηση αυτή δεν θα εφαρμοστεί η διαδικασία Catch ούτε και οι ερωτήσεις με τη γαλάζια κάρτα εξαιτίας της πίεσης χρόνου. Εκ μέρους του Συμβουλίου θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ε, Λιθανικής Προεδρίας, τον κύριο Λασκεβίτσιος, που ομιλεί και εκ μέρους της ΥΠΑ της εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλεια της κυρίας Άστον. Κύριε Λεσκεβίτσιος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Από τη στιγμή που μιλάμε, λαμβάνουν χώρα δραματικά γεγονότα στην πρωτεύουσα του Αιγύπτου, το Κάιρο. Και είναι η στιγμή όπου όλοι εδώ σε αυτό το σώμα θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια έκκληση σε όλα τα μέρη να σταματήσουν την κλιμάκωση της έντασης και τη βία και να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση στην κρίση μέσα από το διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη. Η στιγμή αυτή είναι πολύ κρίσιμη και θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα υπέρ της ε, δημοκρατικής λύσης. Μόνο μια πολιτική ε, διαδικασία που θα οδηγήσει στην επάνωδο της δημοκρατίας θα επιλύσει την τρέχουσα κρίση. Είπα το αντιπρόσωπο και αντιπρόεδρος Άστον έχει παροτρύνει σήμερα το πρωί ε, ε, προς αυτοσυγκράτηση και ζήτησε από όλα τα, μέλη, τα μέρη να βρουν μια πολιτική λύση με βάση ένα ουσιαστικό ε, διάλογο, όπως τόνισε η αντιπροσώπους από την αρχή της Αραβικής Άνοιξης. Η βαθιά δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με εκλογές και πλειοψηφίες, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ε, μια ε, ανεξάρτητη ε, δικαστική, δικαστικό σώμα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την, της ελευθερία της έκφρασης. Η δημοκρατία σημαίνει να αφουγκράζεσαι τους πολίτες και να ακούγονται οι φωνές όλων των ανθρώπων και όχι μόνο της πλειοψηφίας. Εμείς βλέπουμε τις βαθιές ανησυχίες των διαδηλωτών, ε, βλέπουμε την απώλεια ζώων και τον αριθμό των τραυματιών, μεγάλη αριθμή ε, σεξουαλικών κακοποιήσεων γυναικών διαδηλωτών είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Είπα ε, Αντιπρόσωπος ήταν στην Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα και συζήτησε τη κατάσταση με τον Πρόεδρο και την θέση με ένα σαφές μήνυμα έχουμε από την αρχή της Επανάστασης ότι η Επανάσταση ανήκει στους ανθρώπους, στο λαό και θα πρέπει οι προσδοκίες των Αιγυπτίων πολιτών να ικανοποιηθούν μέσα από το διάλογο. Θα συνεχίσουμε σε όλα τα επίπεδα να προσπαθούμε προσπαθήσουμε να βρούμε ε, λύσεις και να εισακουστούν οι φωνές των, του Αιγυπτιακού λαού. μεγαλύτερη πρόκληση για την Αίγυπτο είναι η πόλωση της ε, κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Όπως έχουμε δει, εκατομμύρια διαδηλωτές ε, πλημμύρισαν τους δρόμους της Αιγύπτου και ζήτησαν από τον πρόεδρο Μόρση να αποχωρήσει και ζητούσαν πρόορες εκλογές γίναν και μικρότερες διαδηλώσεις σε άλλα περιφερειακά κέντρα. Μόνο πριν από ένα χρόνο εξελέγει ο Μοχάμετ Μόρση μέσα από τη μουσουλμανική ε, αδελφότητα ως πρόεδρος. Ένα ορόσημο στην μεταβατική περίοδο της Αιγύπτου, το οποίο καλωσόρισε και η διεθνής κοινότητα. Ο πρόεδρος Μόρση αμέσως αυτό ανακηρύχθηκε αντιπρόσωπος όλων των Αιγυπτίων και οργάνωσε το μη στρατιωτικό μέρος ε, των πολιτών. Από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει χρόνο και ε, προσπάθειες ε, να ε, βοηθήσει τη μεταβατική περίοδο στην Αίγυπτο. Ο ειδικός αντιπρόσωπος, ο Μπερναντίνο Λεόν, έκανε αρκετά συζητήσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για να ξεβρεθεί κοινό έδαφος στα πολιτικά και οικονομικά θέματα. Όλοι οι συνομιλητές ε, συμφώνησαν ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει πολιτικά και οικονομικά προβλήματα και όλοι συμφώνησαν ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να το πράξουν και δυστυχώς ο ανασχηματισμός ε, δεν είχε τα αποτελέσματα που επιθυμούσε η χώρα και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πολύ ενεργή στην στήριξη της Αιγύπτου. και η Κάθριν Άστον τόνισε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο. Επίσης ο κύριος Λαμπρίδης μετάβη στο Κάιρο στα μέσα του Ιούνιου και τόνισε την σημασία της οικοδόμησης μιας κοινωνίας με βάση την ενμετάξη και τον σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε ε, τεχνική στήριξη στην σύνταξη νομοθεσίας και στον νόμο κατά της βίας κατά των γενικών. Αυτά αποτελέσματα ε, αυτών των προσπαθειών αποτέλεσαν ε, βοήθησαν την ελληνική πλευρά να συνεργαστεί αυτή για την διατύπωση του ε, νόμου για τις ΜΚΟ. η Αίγυπτος έχει επιβεβαιώσει την βούλησή της να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα, τις άλλες προβληματικές διατάξεις του προσχεδίου του νόμου. Τέλος, σε σχέση με τις ε, καταδίκες των 43 ΜΚΟ, η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι οι Αιγυπτιακές αρχές αναμένουν την πολιτική πολιτικό χρόνο για την ανέβρεση μιας λύσης. Εκτός από το πολιτικό αδιέξοδο, την έλλειψη εμπιστοσύνη ε, που οδήγησε σε αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις και το γεγονός ότι πέσαν πάνω από δύο χρόνια και η Αιγύπτη ε, ε, είναι σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν το 2011. Δυστυχώς η οριστικοποίηση μιας διευθέτησης του ΔΝΤΑΦ συνεχίζεται να αναβάλλεται. Οι δημόσιες υπηρεσίε ε, ε, συνεχώς δυσλειτουργούν, υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. Και ε, η Αίγυπτος προσπαθεί συνεχώς να ολοκληρώσει τη μεταβατική περίοδο αυτή. Αλλά η Αίγυπτος θα πρέπει να βοηθήσει με τη σειρά της. Η Η ποιος χρειάζεται τουρισμό και άμεσες επενδύσεις για να ε, εκπληρώσει τις ε, οικονομικές της δεσμεύσεις και χρειάζεται σταθερότητα και πραγματική προσήλωση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και όπως είπα και στην αρχή η κατάσταση εκεί στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή εξελίσσεται καθώς μιλάμε. Τα γεγονότα είναι πολύ δραματικά και όπως το έθεσα και στην αρχή, ήρθε η στιγμή για όλους να καλέσουμε τα μέρη να αποφύγουν την βία και την κλιμάκωση της έντασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λασκεβίτσιος. Και περνάμε στους ομιλητές εκ μέρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρώτα θα δώσω το λόγο για τρία λεπτά στον κύριο Σαλαφράγκα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Υφυπουργέ, κύριε Γενική Γραμματεύ, κυρίε και κύριοι. Η διαδικασία μετάβαση στην Αίγυπτο περνά από δραματικέ στιγμέ και έχουμε συγκεχημένε ε, ειδήσει για την κατάσταση του Πρόεδρου Μόρση. Πριν από μία ώρα έληξε η προθεσμία που έδωσε ο στρατό στην κυβέρνηση για να ξεπεραστεί η σοβαρή κατάσταση που βιώνει η χώρα και που χαρακτηρίζεται από μια πόλωση, από βία επεισόδια, από απώλεια από ανθρώπινων ζωών, από σύνθεση της κυβέρνησης και μια βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση. Η Αίγυπτος, κύριε Πρόεδρε, από πολιτική, οικονομική και κοινωνική άποψη βρίσκεται σε αδιέξοδο. Βρίσκεται σε μια συμφόρηση. Και ποια, ποιο είναι το μήνυμα που μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να στείλουμε υπό αυτές τις περιστάσεις. Καταρχήν ένα μήνυμα και μια έκκληση για αυτοσυγκράτηση, ε, ηρεμία και διάλογο προκειμένου να υπερκεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Δεύτερον, θα πρέπει να εισακουστεί η φωνή του λαού μέσω ενός διαλόγου που θα περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών και θα την αποκλείει. Είναι αδύνατο να ευοδοθεί μια διαδικασία μετάβασης χωρίς συνένεση και αυτή η συνένεση θα πρέπει να αντανακλάται σε ένα σύνταγμα που θα προβλέπει τη χωρισμό των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά την πρόβλεψη για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και φυσικά σεβασμό των μειονοτήτων. Θα πρέπει να χαραχθεί και ένας οδικός χάρτης μέσω μιας κυβέρνησης εθνικής εμφυλίωσης, μια αναθεώρηση του συντάγματος αλλά και του εκλογικού νόμου προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι ένα σύμβολο στον αραβικό κόσμο και θα είναι και κέρδος παράγοντας στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Μια διαδικασία που κλονίζεται αυτή τη στιγμή από την κατάσταση στη Συρία, από το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν και ως εκ τούτου η Αίγυπτος ε, είναι ένα σημαντικός παράγοντας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να οδηγηθεί σε αστάθεια. Θα πρέπει η Αίγυπτος να δει το δρόμο της να βρει την πορεία της και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, είναι προ... να συνεχίσει να είναι πρόθυμη να προσπίσει, να προσπίσει την ειρήνη, το διάλογο, τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία και την ανάκαμψη της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και για τρία λεπτά επίσης το λόγο έχει η κυρία Δεκεϊζέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει ξεκινήσει η διελκυστίδα μεταξύ της, του στρατού και της κυβέρνησης του κ. Μόρση τη στιγμή που μιλάμε. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, σας, να υπενθυμίσω την υποστήριξή μας προς τον Αιγυπτιακό λαό που το 2011 έδωσε μάχη για περισσότερη ελευθερία, περισσότερη αξιοπρέπεια και φυσικά και μια οικονομική ευημερία. Ο κύριος Μόρση, ο πρόεδρος Μόρση, εξελέγει με δημοκρατικό τρόπο μετά από νομότυπες εκλογές. Δεν κατάφερε όμως να δώσει στον Αιγυπτιακό λαό αυτό που περίμενε και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Βέβαια δεν πρόκειται με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα να βρεθεί η λύση και τη στιγμή που σας μιλώ εγώ, τη στιγμή που ο στρατός αναπτύσσεται στους δρόμους του Καΐρου και έχει καταλάβει το κτίριο της τηλεόρασης, θα ήθελα να απευθύνουμε έκκληση για μια διαδικασία ειρηνικής μετάβασης προς τη δημοκρατία. Και από τη στιγμή που ο πρόεδρος Μόρση εξελέγει ε, νομότυπα, ε, θα πρέπει να, να δούμε πού δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Χάθηκε η κλωστή φαντουργία, ε, χάθηκαν θέσεις απασχόλησης, υποβαθμίστηκε ε, το νόμισμα, υποτιμήθηκε το Αιγυπτιακό νόμισμα. Όλες αυτές οι οικονομικές ε, δυσχέρειες ε, δεν συνέβαλαν συνέβαλε μάλλον στο να μην μπορέσει η Αίγυπτος να πάρει τη βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμηθείτε αυτό το βεβαιασμένο δημοψήφισμα και τι είχαμε πει για τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν εξασφαλίζει τα απαραίτητα δικαιώματα είπαμε και θα συνεχίσουμε να στιγματίζουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ ενισχυτικές και για το μέλλον. Φυσικά το μέλλον θα περάσει από μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και φυσικά θα πρέπει να διεξαχθούν και νέες εκλογές. Αυτό θα το αποφασίσει ο Αιγυπτιακός λαός, αλλά θα πρέπει και οι υποσχέσεις του 2011 και ως προς τη δημοκρατία και ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα να τηρηθούν, γιατί δεν θα έχουμε ειρήνη στην Αίγυπτο και δημοκρατική μετάβαση αν δεν υλοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Η κυρία Αστόν έχει προνομιακή σχέση με την ε, Αιγυπτιακή κυβέρνηση και πέρυσι το Νοέμβριο την περιμέναμε ε, δίπλα στον πρόεδρο Μόρση και στην ε, κυρία Κλίντον. Θέλαμε, θα θέλαμε η κυρία Άστον να χρησιμοποιήσει αυτές τις προνομιούχες σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με την κυβέρνηση Αιγύπτου για να διευκολύνει την ανέβρεση λύσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει τόσο πολλά για τη δημοκρατική μετάβαση στις αραβικές χώρες δεν θα πρέπει στη στιγμή της, ε, τη πιο κέρια στιγμή να επισκιάζεται από άλλους ε, ε, εταίρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει τη δέσμευσή της και να μας δείξει την, τις ικανότητες της κυρία Άστον. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Το λόγο έχει η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ενώ εμείς ε, συζητούμε αυτή τη στιγμή, κατακλείζονται οι δρόμοι στην Αίγυπτο από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν ποτέ σημειωθεί. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να στρέψει τον ένα κατά τον άλλον. Οι ε, βίες συγκρούσεις και ιδιαίτερα αμφίλιος πόλεμος πρέπει να αποφευχθούν. Ο πρόεδρος Μόρση αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση διεδέχεται την ε, διεφθαρμένη κυβέρνηση Μουμπάρακ είχε πολλές ευκαιρίες να μεταρρυθμίσει την οικονομία και να προχωρήσει προς τη δημοκρατία η ποινικοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η αποτυχία να εμποδίσει την άνοδο των τιμών του ψωμιού και των καυσίμων ε, είχαν ως συνέπεια να χάσει την νομιμότητα που είχε στα μάτια πολλών Αιγυπτιών. Και είναι ενθαρρυντικό που βλέπουμε τόσοι πολλοί Αιγύπτιοι να απορρίπτουν τη δικτατορία της πλειοψηφίας και να θέλουν κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα για όλους. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς το να μπορείς να ψηφίζεις. Και η Ένωση πρέπει και αυτή να τα πάει καλύτερα. Μέχρι στιγμής ε, το σύνθημά μας ε, περισσότερα για περισσότερα ακούγεται κενό περιεχομένου. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους στην Αίγυπτο, να βοηθήσουμε για να αποφευχθεί η βία ε, στο άμεσο μέλλον, για να υπάρξει διάλογος χωρίς αξοπλισμούς, ε, χωρίς αποκλεισμούς για να περάσουμε σε μια κοινωνία που να βασίζεται στο κράτος του νόμου, προς την οικονομική ανάκαμψη και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, σεβόμενοι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Αιγυπτίων. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει δημοκρατική προοπτική προς, για τους νέους Αιγυπτίους που είναι τόσο άριθμοι που θέλουν προοπτικές και που προσβλέπουν και κοιτάζουν προς την Ευρώπη. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ασάκε από πλευρά των Πρασίνων. Δύο λεπτά επίση. η συνάδελφο Γιούντιτ ε, ε, Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Μόρση από τότε που ανέλαβε τον καλέσαμε στο σώμα μας αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Και βλέποντας τι έγινε τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι λυπηρό, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί του, όπως συζητήσει που είχαμε χθε με τον Πρωθυπουργό κύριο Όρμπαν. Ο κύριος Μόρση δεν έδειξε και τόσο δημοκρατικά ε, ε, χαρακτηριστικά. Όλο και, περισσότεροι, ε, και και περισσότερο περιοριστικοί νόμοι ψηφίζονταν, για παράδειγμα ο έλεγχο των μη κυβερνικών οργανώσεων, και ε, αναβλήθησαν κάποιες εκλογές. Έχουμε μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Είμαστε εντεθειμένοι να βοηθήσουμε την Αίγυπτο από πλευράς οικονομικής και από πλευράς ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών και ελπίζω ότι δεν είναι σκόπιμο να απελευθερώσουμε τους πόρους που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι για τη βοήθεια. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε προς το παρόν. Μας ε, τρομάζουν αυτά που συμβαίνουν στο Κάιρο πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις για να γίνουν νέες εκλογές, να αναπτυχθεί περισσότερη δημοκρατία, αλλά πρέπει να επιδείξουμε παρουσία. Διότι ξέρετε ότι το δεύτερο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ήταν οι σαλαφιστές. Και ε, ε διερωτώμεθα οι απογοητευμένοι από τον Μόρση προς τα που θα στραφούν. Σίγουρα δεν θα στραφούν όλοι προς την ε, φιλελεύθερη συμμαχία. Πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εξαρτήτων σκεπτομένων, των μειονοτήτων και των γυναικών. Και στην ε, προηγούμενη συζήτηση ε, είπαμε ότι δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω την Αίγυπτο. Δεν θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να σταματήσουμε να απαιτούμε να αναπτυχθεί η δημοκρατία στη χώρα αυτή. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η δημοκρατία είναι ε, δημοκρατία μόνο αν ο πρόεδρος δεν εκλέγεται από το στρατό. Για των, από πλευράς των συντηρητικών δύο λεπτά ο Δόκτωρ Τάνοκ. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ ότι η κατάσταση στην Αίγυπτο ε, είναι ιδιαίτερα σοβαρή και εξελίσσεται από στιγμή σε στιγμή όσο πλησιάζει η προθεσμία που είχε θέσει ο στρατός και ακούσαμε ότι έχουν κατέβει τάγκ στους δρόμους. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα εκατομμύρια των Αιγυπτίων που ποτέ δεν εγκατέλειψαν το όνειρο ελευθερίας, ευημερίας και ασφάλειας όλες τις δεκαετίες της τυραννίας Μουμπάρακ και κατά τον, ε, την Αραβική Άνοιξη και ε, αυτό το χρόνο Τη ε, ε, χαόδους κακοδιαχείρισης του Μόρση που αυτή τη στιγμή αμφισβητείται. Πριν από μερικού μήνε είχα πει ότι οι επαναστάσει είναι με βάση δημοκρατία και όχι πλήρης μεταμορφώσει. Θα έπρεπε βέβαια μετά από τόσε μεγάλες αλλαγέ να περιμένουμε μια περίοδο αστάθεια, αλλά ο πρόεδρος Μόρση ε, απογοήτευσε και τους διεθνείς εταίρους αλλά και το λαό του Βεβαίως η Αιγύπτιοι πολιτικοί ε, δεν είναι αυτοί που θα υποφέρουν. Ε, αυτοί οι οποίοι παίζουν τον κύριο ρόλο είναι τα εκατομμύρια ε, Αιγυπτίων που θέλουν να ζητήσουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερία. Τα συμφέροντα του Μόρση είναι τα συμφέροντα της σεκταριστικής Ισλαμικής αδελφότητας υπό την ε, ηγεσία των οποίων, υπό την ε, κυβέρνηση των οποίων έχει αυξηθεί η ανισότητα, έχουν περιοριστεί τα δικαιώματα των γυναικών, των κοπτών και ορισμένες φορές επιχειρήθηκε μονομερός να αναλάβει αυτό το κόμμα όλες τις μορφές εξουσίας, κάτι που ούτε και ο Μουμπάρακ δεν τόλμησε να επιχειρήσει. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια διακυβέρνηση. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε την ε, προσπάθεια των Ταμαρόντ που προσπαθούν να γίνουν νέες εκλογές. Δεν πρέπει να υπάρξει δικτατορία και οι ε, διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ειρηνικές, ιδιαίτερα λόγω των συγκρούσεων που σημειώθηκαν ε, μεταξύ ε, των ε, υποστηρικτών του Μόρση και των δυνάμεων ασφαλεία χθε βράδυ στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και που είχαν ω αποτέλεσμα 16 νεκρού. Η Αίγυπτος, στην Αίγυπτο αξίζει καλύτερη μοίρα. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Εκ μέρου τη Γκουε τώρα, για 1,5 λεπτό, ο κύριο Βίλι Μέιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι επόμενε ώρε θα είναι αποφασιστική σημασία, πολύ κρίσιμε και πιστεύω ότι το μήνυμά μα θα πρέπει να στραφεί προς τον πρωταγωνιστή αυτών των ορών που είναι ο Αιγυπτιακός λαός. Ε, εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, ε, αναπτύσσεται ο στρατός με τεθωρακισμένα, με τάγκ και ήδη κατέλαβε το κτίριο της τηλεόρασης. Ε, πρέπει να αποφευθεί μια μοιραία εξέλιξη. Επίσης, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στο Φατούχα Αλσίση, τον ε, αρχηγό των ανάπλων δυνάμεων. Κανείς δεν θα πρέπει να ε, τεθεί υπεράνω του Αιγυπτιακού λαού. Επίσης, ε, το αίτημα των ανταρτών Ταμαρόντ που λένε ότι συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια υπογραφές για να οργανωθούν πρόορες προεδρικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη εγγύηση για μία ανέμακτη μετάβαση και η επανάσταση του γιασεμιού και της πλατείας Ταχρήρη ήταν ε, κοινωνική επανάσταση και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ε, η σεκταριστική προσέγγιση ή η θρησκεία ούτε στην επανάσταση του Γεσεμιού ούτε στην, Ταχρήρ, ε, στην πλατεία Ταχρήρ. Επίσης, ο ρόλος που ανέλαβαν οι αδερφοί μουσουλμάνοι. Πιστεύω ότι η θρησκεια ουτε στην επανασταση του Γιασεμιού ουτε στην πλατεια Ταχρήρη. επισης Ένωση ε, έκανε λάθος. Φαίνεται ότι εμείς στηρίζαμε τους αδερφούς μουσουλμάνους, ενώ αυτό που θέλουμε είναι μια συνταγματική διαδικασία που θα, θα διατρανώνει τον κοσμικό χαρακτήρα του, συνταγμα, του συντάγματος που θα εξασφαλίζει την, το σεβασμό όλων των οικουμενικών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της Ομάδας για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, το λόγο έχει ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί μίλησα στον συνήθι πληροφοριοδότη μου που μου με ενημέρωσε ότι είχαν πεθάνει πολύ στο Κάιρο και πριν από μία ώρα είχαν άλλον ένα φίλο στον αραβικό κόσμο στο τηλέφωνο που με ενημέρωσε ότι είχαν συγκλονιστεί ε, με το γεγονό ότι στι στις μαζικές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δυνάμεις ε, της τάξης. Η αστυνομία είναι απούσα και ε, ο στρατός, ούτε ο στρατός δεν είναι εκεί και ανησυχώ όταν τα βλέπω αυτά. Αν δείτε αυτή την περίπλοκη κατάσταση, το ερώτημα που γεννάτε είναι το εξής. Ναι, υπάρχει κριτική, δικαιολογημένη κριτική εναντίον στον κύριο Μόρση αλλά ε, ε, για, να τον καταναγκάσουν να αποχωρήσει από το αξιώμα του. Η, η Αιγυπτιακή Αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πρόγραμμα διάσωσης της χώρας από μια οικονομική καταστροφή προς την οποία οδεύει. Η, το Φιλελεύθερο Κοσμικό Κόμμα, ε, αν δείτε ε, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, Υπάρχουν πολλά κόμματα, σαλαφιστές, ε, φονταμεταλιστές. Ε, αυτή είναι η τελευταία ελπίδα της Αιγύπτου για να αποτρέψει τον ματηρό χάος και μια, ένα βίο εμφύλιο και ε, δεν είναι ενθαρρυντικές οι προοπτικές. Ευχαριστώ. κύριε Μπέντερ. Τώρα έχει για ένα λεπτό ο φίλος Φραντς Ομπερμάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Ομπάμα ε, προτείνει στον Μόρση να ακούσει τους ε, διαδηλωτές. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά τι βοηθάει τους διαδηλωτές αυτό καθόλου. Αυτοί πολεμάνε για την ελευθερία κατά τη δικτατορία της ε, μουσουλμανικής αδελφότητας, κατά μιας κυβερνήσεως που έλαβε τα τελευταία χρόνια ένα δις από την Ένωση για να βελτιωθεί η δημοκρατία και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς είναι δυνατόν ο Φαν Ρόμπεϊ να προτείνει να υποσχεθούμε άλλα 5 δισεκατομμύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. 60% των χρημάτων αυτών πηγαίνουν ε, σε... και εξαφανίζονται σε σκοτεινά κανάλια. Δεν χρειάζονται ε, περαιτέρω χρηματοδότηση από εμά. Παρ' όλα αυτά, εμεί θέλουμε να του τα δώσουμε. θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συνδέσουμε με ε, προϋποθέσεις. Και όποιος ε, δεν τηρήσει προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από εμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπερμάιερ. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον εκπρόσωπο της Λουθανικής Προεδρίας, τον κύριο Λεσκεβίτσιους, για να σχολιάσει τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση που έγινε. Ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη και δυσχερή στιγμή ε, με την Αίγυπτο να αντιμετωπίζει σοβαρότητες προκλήσεις. Οι επόμενες στιγμές θα είναι πραγματικά κρίσιμες και θα πρέπει να στηρίξουμε, όπως είπα, τη θέση μας στις αρχές και τις αξίες μας. Εδώ δεν μιλούμε για τεχνητές προθεσμίες, ούτε μεροληπτούμε υπέρ ε, της μίας ή της άλλης ομάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, έλαβαν μέρος στη συζήτηση, τον κύριο Σαλαφράγκα, την κυρία Τεκάιζερ, την κυρία Σχάκε, την κυρία Μπράτνερ, τον κύριο Τάνοκ, τον κύριο Μάιερ, και τον κύριο Όμπερμαϊερ. Σας διαβεβαιώ ότι η ανάλυση ε, για την κατάσταση και οι απόψεις μας ε, συμπίπτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να συνεχίσει τη δέσμευσή της ε, και το ενδιαφέρον της για την Αίγυπτο που είναι σημαντικό εταίρο. Αλλά σε τελική ανάλυση μόνο ο αιγυπτιακός λαός θα καθορίσει το πεπρωμένο του και την πορεία της χώρας. Και φυσικά οι αιρετοί ε, θα πρέπει να ακούσουν τη φωνή του λαού και να ξεκινήσουν έναν ανοιχτό και ευρύ διάλογο με όλες τις πλευρές. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Αιγύπτου θα είναι η πόλωση και ο διχασμός. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ικανοποίηση των βλέψεων και των προσδοκιών του Αιγυπτιακού λαού μέσω διαλόγου και συμβιβαστικών λύσεων. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για άμεση επιστροφή στη δημοκρατία με διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και τη διεξαγωγή των εκλογών. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις για συμπερίληψή τους στην, σε μια ειρηνική διαδικασία συμφιλίωσης. Και εμείς από πλευράς μας, αλλά και η Πατή Εκπρόσωπος, θα συνεχίσουμε σε όλα τα επίπεδα να διατρανώνουμε ότι θα πρέπει να ακουστεί η φωνή του Αιγυπτιακού λαού και να συνεχιστεί η ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος από το ΕΛΚ, την ΚΟΕ, τους σοσιαλιστές, τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα αυτά θα γίνει αύριο, το μεσημέρι.